Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Να βρεθήκαμε εδώ για μια πολύ σημαντική συνεδρίαση η οποία δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να δουλέψει με πολύ μικρές προθεσμίες. Είναι επίσης σε θέση να μας συγκεντρώσει όλους μαζί και διαφορετικές επιτροπές να συνεργάζονται με εμπιστοσύνη μία στην άλλη. Θέλω εδώ να βεβαιωθώ ότι συμφωνούμε επί της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Το έγγραφο δεν έχει μεταφραστεί στις ε, διάφορες γλώσσες. Έχουμε μονάχα της ε, την αγγλική έκδοση Θεωρώ ότι αυτό αντίκειται στον κανονισμό μας και αναρωτιέμαι αν μπορεί να ψηφιστεί δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Γιατί θεωρώ ότι αυτό αντίκειται προς τον κανονισμό και είναι θέμα ουσίας. Εάν οι δύο αυτές επιτροπές κάνουν την ψηφοφορία αυτή, εγώ θα αρνηθώ να συμμετάσχω σε αυτήν, για λόγους αρχής. Η μετάφραση θα είναι στη διάθεσή σας για την Ολομέλεια. Τα πορτογαλικά έχουν σταλεί στην ομάδα σας, στην ΚΟΕ, οπότε μπορείτε να τη βρείτε εκεί. Όχι, δεν έχουμε τα πορτογαλικά, έχουμε ένα σχέδιο, αλλά δεν έχουμε την πλήρη εκδοχή, ούτε στα πορτογαλικά, ούτε σε καμία άλλη γλώσσα. Πρόεδρος, σας διαβεβαιώνω πάντως ότι οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες για τους ευρωβουλευτές, τις διάφορες γλώσσες δηλαδή, μέχρι την Ολομέλεια. Πριν την Ολομέλεια θα τις έχετε στη διάθεσή σας. Τώρα θέλω να βεβαιωθώ ότι έχετε τα πρακτικά τη συνεδρία στις 20 Απριλίου και ότι το σχέδιο αυτό πρακτικών σας βρίσκει σύμφωνος. Δεν έχετε παρατηρήσεις. Σωστά. Ωραία, 21 Απριλίου θα θυμόσαστε ότι ψηφίσαμε ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό συζητήθηκε σε τριμερή διάλογο επί μακρό. Η συνάντηση εκείνη όμως ήταν καρποφόρα και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε μια διατύπωση που δεν είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που εγκρίναμε τότε και γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία να επαληθεύσουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι δύο επιτροπές μας εγκρίνουν την διατύπωση αυτή στην οποία καταλήξαμε μετά από τον τριμερή διάλογο. Ίσως ο Ρομπέρτο να έχει κάτι να προσθέσει πριν ακούσουμε τους συζητητές και ψηφίσουμε. Ευχαριστώ Ζων. Πριν δώσω το λόγο στους συζητητές θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διαπραγματευτική ομάδα, το προσωπικό, τη γραμματεία, τις πολιτικές ομάδες, γιατί όλοι δούλεψαν σκληρά και πετύχαμε να τηρήσουμε την προθεσμία, που ήταν τόσο μικρή, και να ολοκληρώσουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, τηρώντας πλήρως, θα έλεγα, την εντολή των δύο επιτροπών. Γιατί το τελικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στα πορτογαλικά, έχει σταλεί στα πορτογαλικά, δείχνει ότι πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια επιτυχία στην οποία καταλήξαμε από κοινού. Με καλή συνεργασία μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν και σας ευχαριστώ όλους. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σύντομα στους δύο εισηγητές. Πρώτα ο Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο πρόεδρους να ευχαριστήσω τον ε, συνεισηγητή μου όλ και όλους τους κοιόδης ε, εισηγητές. Βεβαίω ε, ευχαριστώ τις γραμματείες των δύο επιτροπών, καθώς επίσης και τα μέλη των πολιτικών ομάδων, του συμβούλους δηλαδή των πολιτικών ομάδων, Ιδιαίτερο δε τον σύμβουλο του δικού μας ε, κόμματος, ε, κόμμα, συγγνώμη, της δικιάς μου πολιτικής ομάδας, ε, τους δύο συμβούλους μάλιστα, γιατί κάναμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, που όμως δεν είναι ίδιος με αυτή, με αυτή της 20 Απριλίου, γιατί είναι καλύτερη η δουλειά που κάναμε. Έχουμε δηλαδή ένα βελτιωμένο κείμενο σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Στην αρχή το θεωρούσαμε αδύνατο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Μειώσαμε την Connecting Europe Facility και το, Ευρώπη 20, το Ενορίζοντα 2020 σε ένα Συνεχίσαμε την εργασία και την προσπάθεια ε, δώσαμε ε, ε, δημοκρατική νομιμότητα στο Ταμείο, απαιτήσαμε και πετύχαμε διαφάνεια με διάφορους τρόπους καθώς επίσης και με τις διάφορες εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνονται στα τακτά διαθήματα. Εάν ε, δεν λειτουργήσει καλά το Ταμείο, η Κομισιόν ε, οφείλει να κάνει νομοθετική πρόταση βελτίωσης και αν δεν λειτουργήσει καθόλου καλά θα πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι αυτή η πλατφόρμα, η συνοδευτική, η οποία ε, ε, στο 1 της τρίτο αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και βεβαίως οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νέο ταμείο, ένα εργαλείο το οποίο είναι ε, επιπρόσθετο, είναι συμπληρωματικό, θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την, ε, ε, και την απασχόληση και ε, να πω ότι το Κοινοβούλιο συνέβαλε έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν και θα πρέπει να δραχτούμε αυτή της νέας ευκαιρίας που ανοίγεται μπροστά μας για το μέλλον, που όμως ταυτόχρονα αποτελεί και ε, πρόκληση. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το στόχο μας, δηλαδή μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Thank you. Udo Udo ε, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο Προέδρους των Επιτροπών. Εννέα τριμερείς διάλογοι, συχνά μέχρι τα ξημερώματα, ο αποφασιστικός από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί. Πολύ δουλειά και από πλευράς της γραμματείας. Ευχαριστώ τη γραμματεία, ευχαριστώ τους συνεργάτες. Στα γραφεία μας, τις πολιτικές ομάδες αλλά και τους δύο προέδρους των επιτροπών αυτών. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη συνεδρίαση αρνήθηκαν να δώσουν σε μένα και στον ε, Χωσέ Φερνάντη την πιστοτική κάρτα για να επενδύσουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο Χωσέ Μανουέλ Βερνάντη και εγώ λοιπόν ήμασταν ε, τελείως αφελεί. Ε, δεν τολμήσαν να μας δώσουν ε, την πιστοτική του κάρτα. Αλλά σήμερα έχει αλλάξει τελείω η κατάσταση. Σήμερα ψηφίζουν και αυτοί μαζί. Καταφέραμε πάντως κάτι. Καταφέραμε μία τελείω νέα δομή και θα είμαστε συνυπεύθυνοι για τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου θα επηρεάσουν τη λειτουργία του όχι μόνο προς όφελος ε, των ε, δύο πρόεδρων των επιτροπών μας, αλλά ε, προς όφελος των φορολογούμενων και των πολιτών της Ευρώπης. Καταφέραμε να υπάρχουν κριτήρια επενδύσεων για αυτούς που επενδύουν όχι στο χθες αλλά στο αύριο. Προγράμματα για το μέλλον προγράμματα για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με νέους πόρους που έχουμε διασφαλίσει στον κανονισμό. Τα σχετικά κεφάλαια έχουν διατυπωθεί σωστά. Έχουμε κατευθυντήρες γραμμές για τις επενδύσεις. με απόφαση του Κοινοβουλίου έχουμε καταφέρει να συμπεριλαφθεί κάτι το οποίο δεν ήθελαν ε, το, κοινοβούλιο και, ε, ε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αρχικά. Επηρεάζουμε λοιπόν και τον τρόπο που γίνεται η επιλογή των προγραμμάτων με αντικειμενικά κριτήρια χρησιμότητας. Έχουμε διανύσει λοιπόν πολύ δρόμο και όλα αυτά αποτελούν σημαντική επιτυχία. Τα κράτη-μέλη μπορούν και πρέπει να επενδύσουν στο, με, το Ταμείο αυτό. Για να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Η Κομισιόν θα κάνει επίσης τη σχετική δήλωση για να τονίσει ακριβώς αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες διότι έκανε καταπληκτική δουλειά στο ε, θέμα του προϋπολογισμού. Καταφέραμε να πετύχουμε έναν καλό συμβιβασμό πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε να εργαστούμε στο μέλλον και με βάση τον οποίο θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα, τις ελλείψεις που δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτή τη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εισηγητές των δύο επιτροπών, τους σκιώδεις εισηγητές επίσης. Κατά την πρώτη συνεδρίαση είπαμε ότι αν καταφέρουμε από κοινού κάτι, θα γράψει ιστορία το κοινοβούλιο μας ε, ξεπερνώντας τα όρια των πολιτικών ομάδων των επιτροπών και θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε. Έτσι λοιπόν η συνεργασία και η πρόοδος μας οδήγησαν σε επιτυχία και ελπίζω να μπορεί να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία και στο μέλλον σε άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι στους δύο εισηγητές μας. Ζων. Και εγώ φυσικά ε, θέλω να επαναλάβω τη δική μου ικανοποίηση και την ευχαριστία μου για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συνταχθεί στο εγχείρημα αυτό. Ο τελευταίος τρίλογος τελείωσε στις 8 η ώρα το πρωί. Αλλά η σαφήνεια, η αποφασιστικότητα, η επιμονή μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αίσιο πέρας και το κείμενο που έχουμε σήμερα είναι ένα κείμενο το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με αυτό το οποίο είχε εγκριθεί στις 20 Απριλίου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επιτύχουμε μια μεγαλύτερη ε, πλειοψηφία. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στη ψηφοφορία. Έχετε την κάρτα σας. Θα γίνει ονομαστική κλίση. Να κάνουμε πρώτα μία δοκιμή ένα έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για δοκιμαστική ψηφοφορία. Stock taking is not working. So, okay. Δεν λειτουργεί. Everybody has the card. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Δύο μέλη, ένα μέλος χωρίς κάρτα. GUE member, correct? Από την GUE, εντάξει. Now we can proceed. Yeah. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Vous n'avez pas Ψηφίσατε όλοι. Δύο βουλευτέ δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Πέρα τι ψηφοφορίε. 78 ψήφισαν, 63 υπέρ, 14 κατά και μία αποχή. Και αυτός που δεν είχε την κάρτα του, κατά, καταψήφισε. 15 ψήφι κατά. Μα νομίζω ότι μπορούμε να συγχαρούμε τους δύο εισηγητές. Ο κύριος Κάρας. Η κάρτα μου δεν δούλεψε. Μια ψηφο ακόμα υπέρ. 79 με 15. 64 με 15. Η επόμενη λοιπόν. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην επόμενη μήνυ Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτοιμη να συζητήσει μαζί μας για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρία. Σα ευχαριστώ.